Λοιπόν, ξεκινάμε. Η ημερήσια διάταξη ε, μπορεί να εγκριθεί εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 15 η Οκτωβρίου μπορεί να εγκριθεί αν δεν υπάρχουν ενστάσεις. Ανακοίνωση της Προέδρου. Ανακοινώσεις Προέδρου δεν υπάρχουν. Σήμερα έχουμε την πρόθεση να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εάν μου επιτρέπετε θα διατυπώσω ένα αίτημα όσον αφορά την προσεχή ημερήσια διάταξη τη Επιτροπής μας. Θα ήθελα να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη ένα σημείο όσον αφορά την εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση σε σχέση με το πακέτο για την κινητικότητα. Στην ε, ε, Επιτροπή δεν έχει γίνει συζήτηση ε, για το θέμα αυτό ε, λυπούμε για το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις και για το γεγονός ότι ορισμένοι μη βουλευτές έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κείμενα των συμβαστικών προτάσεων. Ε, θα πρότεινα λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται υπό εξέλιξη. Ε, ευχαριστώ πολύ, θα το σημειώσω και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την κατάσταση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από, την, ε, από το πρόγραμμα InvestEU. Ε, καταρχήν, θα πρέπει να δούμε αν έχουμε απαρτία. Θα κάνουμε μία ε, ηλεκτρονική δοκιμή. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Κύριε Πίπερ, δεν, χρειάζεται να ψηφίσετε. Είναι καλός ο αριθμός των ψήφων, ακόμα και για το ΕΛΚ. Αρκεί. Ωραία λοιπόν. Υπάρχει απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση Βάντε για την πρόταση κανονισμού σε σχέση με το πρόγραμμα InvestEU. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σεβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε. Η 69 παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας για την 69 απορρίπτεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται περνάμε άμεσα στην 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Οχ, ε, όχι, 80 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα γίνει παλήθευση. Για την 80 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα πάμε στη συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική α5 υπέρ κατά αποχές θα γίνει ηλεκτρονική υπαλήθευση για την τροπολογία για τη συνδυστικη μαλλον μάλλον 5α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5β. Α. Ε, συγγνώμη. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απο, ε, εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα περάσουμε τώρα στη τροπολογία υπαριθμών 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ, Θέλετε να γίνει επελήθευση. Επελήθευση για την 135 της κυρίας Ρουβόνταλόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δυστυχώς Απορρίπτεται. Θα συνεχίσουμε. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επαλήθευση. Ωραία. Λοιπόν, για την 136 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 136 εγκρίνεται. Να με εμπιστεύεστε παρακαλώ. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 επαλήθευση 138 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται δυστυχώς 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139. Επαλήθευση. Πέρασε ψηφοφορίες. Α, απορρίπτεται. Συνεχίζουν. 140 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά, υπέρ, κατά, αποχές, απο... εγκρίνεται. Για την 149. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. 149. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 153 και 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας. Ε, τι έγινε εδώ. Θα συνεχίσουμε, δεν ε, διασκεδάζουμε εδώ, δεν παίζουμε. 155 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 156 ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στο 162 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 161 μάλλον. Α, όχι, 171, συγγνώμη. Μα τι γίνεται εδώ. 20. Πρέπει να αλλάξω φακούς. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 174 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 και 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 177 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική υπαριθμών 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ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 αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33. Α, 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Συγγνώμη, 39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επαλήθευση για τη 49 παρακαλώ Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται συνεπώς. 14 συμβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση για την 54, παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση για την 57. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Πέρας της ψηφοφορίας. Όχι, απορρίπτεται. Καλώ ε, καλώς επαληθεύσαμε. 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι ξεκάθαρο. Για την 61 παρακαλώ να γίνει επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά αποχές, δεν είναι ξεκάθαρο. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 63 άρχεται η ψηφοφορία. πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα γίνει επαλήθευση κύριε Ντέλη. Παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας Απορρίπτεται 65-66 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία, ωραία επαλήθηση είναι 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα της έκθεσης παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Υπέρ 29 κατά 13 ε, η έκθεση εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Και συνεχίζουμε. Nous passons désormais à la proposition de règlement. Περνάμε στην πρόταση κανονισμού θέσπιση του προγράμματος για την ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027. Η κυρία Κλούνα είναι η συγγήτρια. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 89 υπέρ. block vote. Δηλαδή, παρνάμε κατευθείαν ε, στην 91. Γιατί απορρίφθηκε η 88. 91 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές. Έλκ τι κάνετε. Ξαναρχίσουμε. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ Κύριε Κράμερ, θέλετε παλήθευση για ποια. Την 97. Θέλετε να επαληθεύσουμε την 97. Ψηφίζουμε για την 97, παρακαλώ. Αμαμό 97. 97. Allez, je ferme le vote, amendement 4. Λήξη. Απορρίπτεται. Εδώ είμαστε για να ελέγχουμε. Κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, υπήρχε πρόβλημα στη μετάφραση. Συνεχίζουμε. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπάρχει ένα θόρυβος ε, 107 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε. 625 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 Allez, je Πέρας. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 και 42 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνονται. 43 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο. Θέλετε να επαληθεύσουμε την 53. Μάλιστα, για την 53 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Ψηφίσατε όλοι. Allez, c'est bon. Je ferme le vote. Plus 40... Υπέρ 45, 2 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται η έκθεση της κυρίας Κλούν. Et nous continuons, s'il vous plaît. Και συνεχίζουμε. Avec Madame Virkunen, votre rapport με την έκθεση της κυρίας Βιρκούνεν. Το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη για την έρευνα. Καλημέρα, Ντομινίκ. <laughs> Allons-y. C'est le rapport de Madame Virkunen. Amendement 38, qui est pour? 38, υπέρ, κατά. Αποχές, Γκρίνεται. 39, υπέρ,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 αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να επαληθεύσουμε τη 49 49 πέρας Γκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54. Θέλετε να επαληθεύσουμε την 53. Έχουμε μία παραπάνω ψήφο από το ΕΛΚ. Κάποιος ψήφισε που δεν έπρεπε. Υποσύρουμε την κάρτα, ωραία. Λήξη. Απορρίπτεται 53. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ποια θέλετε να επελθεύσουμε. Την 90. Ψηφίζουμε την 90. Je ferme le... Allez. Il y en a un encore de trop. Hein. Άλλοι έχουμε έναν παραπάνω. Allez, je ferme le vote. Λήξη. Απορρίπτεται. Και 91 απορρίπτεται, 92. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτω. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτω. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτωται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 94. το έλεγχο, οι σοσιαλιστές θέλουν έλεγχο. Λήξη. Απορρίπτεται. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 96. Je ferme le vote et c'est rejeté. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 98. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ Κύριε Μαρινέσκου ήρθατε Άρχεται η ψηφοφορία για την 100 Πέρας για την 100. Απορρίπτεται κύριε Βερτρέσκου, λυπάμαι. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. συγκρίνεται. 104. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 ναι στην 105 είμαστε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές. Α, 9, 9, διορθώνει η πρόεδρος, ξαναρχίζουμε. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την τροπολογία Μαρινέσκου. Πέρας. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε τη 10. Και Απορρίπτεται. Ένα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στη 12 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. και περνάμε συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Περνάμε στην 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 για την 35 να ελέγξουμε παρακαλώ. 35. Λήξη. Και απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Πέρας. 44 υπέρ 2 κατά 2 αποχές. Κυρία Βερκούνεν, εγκρίνεται. Μπράβο σας. Allez, nous continuons toujours avec vous, Madame Virkunen. Συνεχίζουμε με εσάς, κυρία Βερκούνεν, για το πρόγραμμα έρευνας. Πάλι ορίζουν Ευρώπη.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 56 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 58 καταπίπτει 59 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Λοιπόν, συνεχίζουμε να ελπίζουμε. 68. Υπέρ, κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Για να ψηφίσουμε την 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Je ferme le vote. Λήξη. Εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 να επαληθεύσουμε την 69. Je 6 για την 69 απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται για να ελέγξουμε την 72. Λήξη. Απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 97 ως 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106. Θέλετε έλεγχο. Να ψηφίσουμε την 105 παρακαλώ. Λήξη. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερις ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάλι τέσσερις ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε για την 125 άρχεται η ψηφοφορία. Je vais fermer le vote. Λήξη. Εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνονται. 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. C'est trop pour Marinescu. Allez, on continue. 135, qui est pour κατά, εποχές, εγκρίνεται. Trois amendements Τρεις καταπίπτουν. Συμβαστική 8 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 140 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές γκρίνεται. Τρει ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρεις ταυτόσημες υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνονται. Δύο ταυτόσημες υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνονται. 159 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τρεις ταυτόσημες υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνονται. Ακόμα τρεις υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνονται. 166 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 167 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 169 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές,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 Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην ψηφοφορία του συνόλου του κειμένου ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Allez, je ferme le pot. Λήξη. 44. 44 υπέρ, 2 αποχές, 2 κατά. Συγχαρητήρια κυρία Βυρκούνεν, μπράβο σας. Allez, nous continuons, nous continuons. Allez, monsieur, le rapport de monsieur... Λοιπόν, η επόμενη έκθεση που αφορά την ε, Ευρωμεσογειακή Συμφωνία. Α, Έχουμε μία και μόνο ψηφοφορία εδώ. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Allez, je Λήξη. Ψηφίσατε όλοι. 47. 47 υπέρ, μόνο μία αποχή. Συγχαρητήρια στον συγητή. nous continuons avec le rapport de Monsieur Zlotowski concernant les fonds européens de développement. Έκθεση Zlotowski για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις. Είστε έτοιμοι. Συμβαστική είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά συμβαστική εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να γίνει επαλήθευση. 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Με μία ψήφο κατά. Παρά, πάνω. 38 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται.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 εγκρίνεται 45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται Μπλοκ Α ε, υπέρ αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να γίνει επαλήθευση για το σύνολο των τροπολογιών από το 50 και μέχρι και την 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. 55 ε, υπέρ κατά δεν είναι ξεκάθαρο για την 55 παλήθευση παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμόν 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, επαλήθευση για την 79, παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 80. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημαστική 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 83. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 84. Ε, Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα 89. Ε, 99, συγγνώμη, εγκρίνεται. 100 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δύο ταυτόσιμες ε, ε, τροπολογίες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 104. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 105 υπέρ, κατά, αποχές, Επαλήθευση για την 105. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107. Επαλήθευση για την 106 παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 108. Για να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαντεκόμπτ, Η 107 έρχεται ψηφοφορία, επαλήθευση. Νομίζω ότι έχει την ίδια πλειοψηφία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες 23 ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ, επαλήθευση για την 109 Πέρα στις ψηφοφορίες είναι η ίδια πλειοψηφία Ντομινίκ. Εκατόν δέκα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ωραία λοιπόν, επαλήφευση για την 110. Πέρας της ψηφοφορίας νομίζω ότι απορρίπτεται. Ωραία επαλήθευση. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112. Θες να γίνει επαλήθευση. Ωραία, 111 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 113 υπέρ. Εκατόν δώδεκα. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές. Τι γίνεται εκεί. Δεν σηκώνεται το χέρι. 113. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Θέλετε να γίνει επαλήθευση. Άντε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 29 ψήφοι περ. Είναι ορισμένοι δεν εμπιστεύονται την πρόεδρό τους, βλέπω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συμβαστική υπαριθμών 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. εγκρίνεται. Ποιος είπε για έλεγχο. Κυρία Βερκούνεν, θέλετε να γίνει επαλήθευση. Ωραία. Πάμε. Για την συμβαστική 6. Λήξη της ψηφοφορίας. 33 ψήφοι υπέρ, 10 ψήφοι κατά, εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην 128 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129. Παληθεύουμε. Πέρα στις ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μπλοκ Β, δύο ταυτόσιμες ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία υπαριθμών 140 ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ. Θέλετε να γίνει επελήθευση για την 145, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. για την 144 υπέρ. Α, εγκρίνεται με μία ψήφο υπέρ παραπάνω. 145. 145 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 151. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 153 <coughs> υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ, συμβιβαστική 9 λέει πρόεδρος, υπέρ, κα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα γίνει επαλήθευση για τη συμβαστική μόνο 9, άρχια την ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές δεν είναι ξεκάθαρο. Θα ήθελα να επαληθευτεί ηλεκτρονικά το 2. Η 2. Πέρας της ψηφοφορίας έχει εγκριθεί. Δεν είναι ξεκάθαρο. 24 υπέρ κατά αποχές. Θα επαληθεύσουμε, κυρία Γκραπίνη. Για την 24 πέρας της ψηφοφορίας έχει απορριφθεί 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές Θέλετε να γίνει επαλήθευση για την 28. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Το σύνολο του κειμένου άρχεται η ψηφοφορία. Η έκθεση λοιπόν του κυρίου Ζλωτόφσκι τίθεται θέση ψηφοφορία, πέρα τη ψηφοφορία. 34 ψήφοι υπέρ, 9 ψήφοι κατά Κύριε Ζλωτόφσκι η έκθεσή σας εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Τελευταία έκθεση της ε, κυρίας Κριστίν Ρεβόλντελό, πρόταση συστατικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι, κυρία Συγήτρια. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε πολλέ τροπολογίε σε μπλοκ. Από τη 12 μέχρι τη 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 79 του κυρίου Μαρινέσκου, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο, μάλιστα. But... Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική τρία, υπέρ. Κατά εποχές. Συγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά Εποχέ, απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Την 89. Πέρας. Et c'est rejeté. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές γκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 108 Υπέρ. Θέλετε έλεγχο της 107. Ψηφίζουμε την 107. Λήξη. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Να επαληθεύσουμε την 114. Λήξη. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται πολλές τροπολογίες μπορούν να συνδυαστούν από την 1 μέχρι την 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Vous voulez 33 Allez, on y Θέλετε να παληθεύσουμε 33, παρακαλώ. Et je vais fermer le Απορρίπτεται, έχετε δίκιο. 34, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάλι πολλές τροπολογίες μαζί μπορούν να συνδυαστούν μέχρι Α, θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες ξεχωριστά μία προς μία. 35, περ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση, μάλιστα για την 35. Allez, j'ouvre le vote. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Έχετε δίκιο, απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. Τριάντα εννιά υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Σαράντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σαράντα ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα θέσουμε το κείμενο στο σύνολό του ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Et Λήξη. 38 υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Συγήτρια, υιοθετείτε η γνωμοδότησή σας, αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε και μισή ώρα νωρίτερα. Μπράβο σας, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Vous avez le droit de me payer un café. Μπορείτε να με κεράσετε ένα καφέ. You are a great chair. Thank you. Uh, I will uh, try to uh, get transferred from Libya to you. Okay, great. C'est envoyé, effectivement.